δυνατότητες πάνω από 22.000 μαθητών που θα αυξάνονται όλο και περισσότερο. Έκλεισε η συζήτηση, κύριε Επίτροπε, και θα ψηφίσουμε αύριο επίσης στις 12.30. Και πάμε στο τελικό σημείο της ημερησίας διάταξης, που είναι η έκθεση του κύριου Τόιρερ για την μελλοντική πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και εσείς κύριε Επίτροπε. Απόψε συζητούμε αργά βέβαια το θέμα αυτό, το οποίο έχει μεγάλη σημασία στο κάτω της γραφής η διαθωτική πολιτική καταλαμβάνει το 37% του ευρωπαϊκού προπολογισμού και ε, σήμερα στα μέσα του 2011 πόσα κονδύλια έχουν απορροφηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία. Δυστυχώ διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένε χώρε μέλη η ικανότητα απορρόφηση υπολείπεται κατά πολύ απέναντι στα όσα κονδύλια θα έπρεπε ήδη να είχαν ε, απορροφηθεί. Νέε χώρε μέλη όπω Βουλγαρία και Ρουμανία δεν τα καταφέρουν καλά. Όχι όμω μόνο οι νέε χώρε μέλη. Και χώρε οι οποίε από πολλά χρόνια και ιδρυτικέ μάλιστα χώρε όπω ε, η Ιταλία, η Καλαβρία για παράδειγμα, 7% λέει η έκθεση των ελεγκτών. Άρα υπολείπεται τεραστίως. Γιατί οι περιφέρειες αυτές δεν μπορούν να απορροφήσουν τα κονδύλια που δίνουμε. Άλλο παράδειγμα βεβαίω η Ελλάδα. Εδώ και πολλούς μήνες έχουμε τονίσει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει τα κονδύλια αυτά και είμαστε ικανοποιημένοι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αρχικώς δεν είχε δώσει σημασία τώρα πλέον αποδίδει μεγάλη σημασία. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ειδικά για την Ελλάδα τόνισε ότι 15 δισεκατομμύρια από τα 20 δεν έχουν διατεθεί. Ο Επίτροπος κ. Χάν πήγε επί τόπου και σκέπτεται τώρα τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθούν οι περιφέρειες αυτές. Πρώτα-πρώτα τίθεται το θέμα της συγχρηματοδότησης ότι βεβαίως οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν τώρα δυσκολίες εν μέση παγκοσμία κρίση να απορροφήσουν τα κονδύλια ειδικότερα για χώρες όπως η Ελλάδα η οποία φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε φάση πάυσης πληρωμών βεβαίως πρέπει να βοηθήσουμε δεν λέω όχι αλλά η συγχρηματοδότηση φαίνεται πως δεν είναι η μοναδική αιτία διότι στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλες περιφέρειες οι οποίες δεν επιθυμούν καν αύξηση της υποστήριξης της συγχρηματοδοτικής υποστήριξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευχαριστημένες με το 80% και θέλουν περισσότερα έργα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί και ποικίλοι λόγοι. Οι διαδικασίες είναι υπερβολικά περίπλοκες. Θα πρέπει να απλουστευτούν. Σε ορισμένες χώρες μέλη οι κεντρικές διοικήσεις των κυβερνήσεων, στις πρωτεύουσες δηλαδή, χρειάζονται υπερβολικά πολύ χρόνο οι δε τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν έχουν αρκετή αποφασιστική αρμοδιότητα για να μπορούν να διαθέτουν τα κονδύλια. Παράδειγμα, ορισμένες περιφέρειες στη Ρουμανία, όπου σε ορισμένες κοινότητες προχωρούν οι αιτήσει σε 20 έως 30 μέρες, στις περιφερειακές διοικήσεις σε 60 μέρες, ενώ οι κεντρικές διοικήσεις χρειάζονται σχεδόν ένα χρόνο. Αυτά είναι λοιπόν ε, ε, περιπτώσεις που δείχνουν ότι πρέπει να γίνει μια μετακύληση της ευθύνης, της αρμοδιότητας από τα πάνω προς τα κάτω. Πού βρίσκεται σήμερα το Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Βαν Ρομπόι, ζήτησε και έλαβε το λόγο για άλλα θέματα. Εδώ μιλούμε για το 37% του συνολικού προϋπολογισμού. 250 δισεκατομμύρια καθυστερούν και δεν απορροφώνται. Θα μπορούσε και η Πολωνική Προεδρία να έχει κάνει προτάσεις, διότι η Πολωνία έχει αποδείξει ότι μπορεί να αυξηθεί η απορροφητικότητα. Υπάρχουν και παραδείγματα λοιπόν της λεγόμενης καλής διακυβέρνησης. Το ίδιο η Εσθονία. Εμείς ως Ευρωβουλή θεωρούμε ότι οι χώρες μέλη είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες, ώστε τα κονδύλια που εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο δίνουμε, εγκρίνουμε υπέρ των πολιτών να φτάσουν στους τελικούς απολύπτες έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να στεθεροποιηθεί η απασχόληση και εδώ αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει την αποφασισμένη πορεία και να ζητήσει από τις χώρες μέλη να οδηγήσουν το, τις προσπάθειες αυτές σε αίσιον πέρας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έκανα την γνωμοδότηση από την Επιτροπή Απαγόρευση και θα ήθελα να χαιρετήσω την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον εισηγητή του, ο οποίο στόχο ήταν να εξετάσει την πολιτική συνοχή από διάφορε ε, οπτικές γωνίες και πώς μπορούμε να ε, κάνουμε καλύτερη χρησιμοποίηση των κονδυλίων, πώς μπορούμε να καταρρύψουμε τα εμπόδια ώστε να υπάρξει καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης των κοινωτικών κονδυλίων από τα κράτη-μέλη. Για μας ε, στην Επιτροπή Επασχόληση είπαμε ότι το πιο σημαντικό ταμείο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που αυτή τη στιγμή τη οικονομική κρίση είναι πολύ σημαντικό, διότι η μείωση των θέσεων απασχόληση είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταλεπινθεί. Ο εισηγητή νομίζω ότι σωστά ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα με την συγχρηματοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εξαιτία των ε, ε, περιορισμών στον προπολογισμό και τις πολιτικές λιτότητε των κρατών μελών. Έτσι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ε, αρκετά ε, ε, χρήματα και δεν μπορούν να υπάρξει χρηματοδότηση και εκ μέρους και για τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι πάρα πολύ αργά, αλλά το θέμα που συζητούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για βελτίωση της απορρόφησης των Ταμείων Συνοχής και των Κοινωνικών Ταμείων για να έχουμε πολύ καλύτερη συνεισφορά των πόρων που έχουμε για την περιφερειακή πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει να δούμε από πού προέρχονται τα προβλήματα απορρότησης και να απλοποιήσουμε τις κανόνες και τις διαδικασίες πρόσβαση όλων των επιχειρημανιών στα κοινωνικά ταμεία και η καλή διαχείρισή τους από τις ε, διοικητικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη και να προωθήσουμε μεγαλύτερη συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των κονδυλίων, των ταμείων. Θα ήθελα ιδιαίτερο να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί όσον αφορά την διχείριση των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ε, ε, υποπασχόλησης εξαιρετίας των οικονομικών προβλήματων. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε στο ευρωπαϊκό ε, σχέδιό μας τον κατάλληλο Δρόμο. Αλλά χρειαζόμαστε καλές πολιτικές και φιλοδοξία για να το επιτύχουμε. Ευχαριστώ κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο στόχος της απορρόφησης της ε, οικονομικής βοήθειας απαιτεί συνεχή προσπάθεια από τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό φυσικά σε αυτό να εμπλακούν και οι τοπικές ε, και περιφερειακές ε, αρχές. Οι κανόνες για αυτά τα κονδύλια είναι πάρα πολύ περίπλοκοι και μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες και λάθη. Και τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειές τους σπαταλούν πολύ χρόνο ε, προσπαθώντας να χειριστούν αυτές τις δυσκολίες. Χρειαζόμαστε κανόνες και διαδικασίες απλούστερες σε όλα τα επίπεδα, ούτω ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια και να γίνεται και καλή διαχείρισή του, χωρί να δημιουργούμε μεγάλε δυσκολίε για του δικαιούχου. Η απλούστευση θα οδηγήσει σε γρήγορη ε, απορρόφηση, υψηλότερα επίπεδα απορρόφησης, ε, λιγότερα λάθη στις αιτήσει και λιγότερες ε, βραχύτερες δηλαδή στην καταβολή των κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των εμπλεκομένων. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ. Η πολιτική συνοχή μας ε, εξασφαλίζει την ε, μείωση των ε, χασμάτων μεταξύ των περιοχών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Εμείς έχουμε χαμηλά ποσοστά απορρόφησης στη Ρουμανία, αλλά την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να μειωθούν τα κονδύλια ε, στα οποία έχει πρόσβαση η Ρουμανία, τα οποία τα χρειάζεται. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για να οργανώσουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα και να τα συντάξουμε εν ευθέτω χρόνο. Χρειαζόμαστε αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για να αναπτύξουμε την ενεργειακή υποδομή και να είμαστε πιο αποδοτικοί σε ό,τι αφορά την ενέργεια ε, στα κτίρια μας. Η Κομισιόν επίσης θα δώσει λεφτά για τις ε, υποδομές των μεταφορών που ανήκουν στις περιοχές σύγκλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές μεταφορές. Θέλω να κρατήσουμε τα κονδύλια χωρίς περικοπές. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχίζοντας, επιτρέψτε, αρχίζοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, δημιουργία Υπουργείου Ευρωπαϊκών Κονδυλίων που θα διαχειριστεί όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε όλους τους τομείς. Αυτή τη στιγμή η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν πρόβλημα απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, κυρίως αυτών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να σας πω ότι εφέτος τον Ιούνιο σταμάτησε τις πληρωμές η Επιτροπή για το δεύτερο περιφερειακό πρόβλημα στη χώρα μας. Και αυτό οφείλεται στα προβλήματα που υπάρχουν με την, ε, δημόσιους που γίνονται για την διανομή αυτών των ε, κονδυλίων. Αυτά τα κονδύλια όμως είναι μια εγγύαση κατά των ε, οικονομικών ανισοτήτων που έχουμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Πιστεύω ότι αν υπάρχει και περιφερειακή ανάπτυξη των δεχτή κρανόμετρων, η απορροφητικότητα των κονδυλίων αυτών των ταμείων θα βελτιωθεί. Στο το 2012 είναι για μας πάρα πολύ αφασιστικό για την εφαρμογή προγραμμάτων με χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο το ποσοστό απορρόφησης από το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθωτικά Ταμεία δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένες χώρες γιατί είναι πολύ χαμηλό, ε, γίνονται πάρα πολλά λάθη και πολλές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν αυτές οι χώρες. Ο χρόνος που ξοδεύουμε για να ψάχνουμε τα λάθη είναι τρομερά μεγάλος. Γι' αυτό θα πρέπει να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του συστήματος. Κάτι άλλο που θα πρέπει να μας ασχολήσει είναι να δούμε γιατί οι προϋποθέσεις δεν γίνονται σεβαστές. Θα ήθελα να σας προτείνω ότι όταν υπάρχουν επίσημα λάθη θα πρέπει να γίνεται ε, μια βαθμολόγηση των συμμετεχόντων ανάλογα με το λάθος που έχουν κάνει. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ακυρώσουμε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε να γίνονται αυτά τα λάθη δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με μικρολάθη, θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα βασικά θέματα. Πρέπει να δούμε όλο το θέμα από μια νέα οπτική γωνία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τόιερ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στη Ρουμανία με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ρουμανία έχει πρόβλημα με την απορρόφηση των κοινωτικών κονδυλίων. Και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση υιοθέτησε μία σειρά μέτρων που κατέληξαν, όπως ελέγχθη, στη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο, με υπουργό τον πρώην Επίτροπο Όρμπαν. Έχουμε Λοιπόν, ελπίδες για την ε, υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων και σήμερα πρέπει να σας πω ότι λάβαμε μία ανακοίνωση από την Επιτροπή σύμφωνα με την οποία δύο από τα δικά μας σχέδια, σχέδια που υποβάλαμε αξίας 720 εκατομμυρίων ευρώ ενεκρίθησαν για δύο project επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Νικολάσετς. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Κομισιόν, μια αποτελεσματική πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν όλες οι περιφέρειες της ευρωπαϊκής ένωσης, γιατί ακυρώνει τις διαφορές και τα χάσματα που υπάρχουν. Το ποσοστό απορρόφησης ε, και η αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων των ε, ταμείων διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια δυστυχώς οι πιο προβληματικές περιφέρειες που χρειάζονται πραγματικά τα κονδύλια απεγνωσμένα καθυστερούν στην απορρόφηση λόγω ε, έλλειψης πόρων από τη συγχρηματοδότηση αλλά και λόγω του ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι και διοικητική υποστήριξη. Θα πρέπει να δοθεί τέτοια διοικητική υποστήριξη ε, σε περιφερειακό επίπεδο με επικεντρωμένο τρόπο. Οι αρχές επίσης θα πρέπει να προσλαμβάνουν προσωπικό πραγματικά καταρτισμένο. Πολλά κράτη έδειξαν ότι όλο και περισσότερο ξοδεύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κονδύλια της Ευρώπης. Ε, η δική μου χώρα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Επίτροπος Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Τόερερ που έθεσε επιτάπητος το σημαντικό αυτό θέμα. Όντως, χρειάζεται να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια, διότι είναι σημαντικά και θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικά στα πλαίσια των επικειμένων συζητήσεων για το μέλλον του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την σύνταξη της εκθέσεως, την οποία θεωρούμε ως σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην συζήτηση για την βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης και υποστήριξη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας ικανοποιεί επίσης ότι η έκθεση αναφέρεται στην απορροφητικότητα, στην ικανότητα απορρόφησης, χρησιμοποιώντας μια ευρύτερη προσέγγιση και ευρύτερες έννοιες της ικανότητας απορρόφησης, πέραν δηλαδή των καθαρά οικονομικών ενιών. Έχει σχέση και με την βελτίωση της χρήσης των κονδυλίων χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο δηλαδή οι πόροι. Η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει κοινό έδαφος για τις αναλύσεις ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν έδειξε την διάθεσή της να υποβάλει τα διαθέσιμα δεδομένα για την ικανότητα απορρόφησης, παρόλο που ορισμένα από αυτά προέρχονται από τις ίδιες τις χώρες μέλη. Μας ανησυχούν και μας οι καθυστερήσεις στην απορροφητικότητα και επίσης οι για τις εκτιμήσεις προσαρμογής ή συμμόρφωσης και για την περίοδο 2007 έως 2013. Η απορρόφηση, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, έχει ωστόσο επιταχυνθεί και ο μέσος όρος είναι στο 29,2% που δείχνει ότι η απορρόφηση κονδυλίων των διαθωτικών ταμείων έχει βελτιωθεί. Από όλες όμως τις παρεμβάσεις που ακούσαμε απόψε είναι σαφές ότι χρειάζεται να διδαχθούμε από την παρούσα περίοδο να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονται οι κανόνες για, τη μελλοντική, για τις μελλοντικές δαπάνες και ενώ τώρα προχωρούμε στην σύνταξη των προτάσεων για την περίοδο 2014 έως 20 θα λάβουμε βεβαίω υπόψη μας όλα αυτά τα διδάγματα. Στις προτάσεις μας θα ενσωματώσουμε και τα αποτελέσματα των αναλύσεων και επίσης ένα σημαντικό μέρος θα είναι και η όθηση και πίεση για μια απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας και στο ευρωπαϊκό αλλά και στο εθνικό επίπεδο. Και εδώ θα πολύ συχνά οι δυσκολίες εμφανίζονται στο τέλος των διαδικασιών. Θα ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να βελτιώσουν την διοικητική τους ικανότητα καθώς και την αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών διότι βλέπουμε συχνά σε ορισμένες χώρες μέλη μια πτώση της διοικητική του ικανότητας και αυτό βέβαια συνεπάγεται μείωση και της ικανότητας απορρόφησης. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε την ιδέα των συνεργασιών και πολυεπιπέδων συνεργασιών των κυβερνήσεων αλλά και συνεργασίες μεταξύ κομισιών και χωρών μελών σε μια προσπάθεια βελτίωσης και της διαχείρισης των ταμείων στο μέλλον. Για να απαντήσω στην κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων υπέρ των Ρώμα, εμείς αναμένουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανυπομονησία μάλιστα, τις εθνικές στρατηγικές που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί τα τέλη του έτους. Μόλις θα τις λάβουμε, θα τις αξιολογήσουμε και θα ξεκινήσουμε μια ευρεία συζήτηση για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά για την ενσωμάτωση των Ρώμα. έκλεισε συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30 αύριο στις 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 και από τις 3 έως τις 9